Καλά σας απόγευμα συνάδελφοι. Προτείνω να αρχίσουμε την ε, απόψινή συζήτηση. Με χαρά υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας της Εστονίας, τον κύριο Σινόφσκι, ο οποίος βρίσκεται εδώ λόγω εστονικής Προεδρίας. Έχουμε πολλά θέματα ενδιαφέροντος, κοινού ενδιαφέροντος και νομίζω ότι θα μπορέσετε να προωθήσετε κατά την Εστονική Προεδρία και έχετε πολλές φιλοδοξίες στον τομέα της υγείας μέσα στα πλαίσια της Προεδρίας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες για το επόμενο εξάμεινο, για το τρέχον εξάμεινο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Εστονικής Προεδρίας στον τομέα της υγείας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαλτέζικη Προεδρία για την εξαιρετική της εργασία κατά τους ε, προηγούμενους έξι μήνες, όπως ξέρετε, από την 1η Ιουλίου έχουμε αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά και την αναλαμβάνουμε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά και βεβαίως με αίσθημα ευθύνης. Ε, το γνωμικό, μάλλον η σκέψη που μας διατρέχει, είναι η ενότητα μέσω της ισορροπίας και εξισορρόπησης θα πρέπει να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες και η υγεία είναι κάτι που μας αφορά άμεσα και ατομικά. Θέλουμε να ζούμε μια υγιή ζωή όλοι οι άνθρωποι έτσι ώστε όλοι μας να μπορούμε να συνεισφέρουμε στην κοινωνία και την οικονομία. Επίσης, σύμφωνα με το, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι Ευρωπαίοι θεωρούν την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, το τέταρτο πιο σημαντικό θέμα στη χώρα τους, βεβαίως μετά από την τρομοκρατία, ανεργία, μετανάστευση και οικονομική κατάσταση. Όπως γνωρίζουμε, ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε χρόνιες ασθένειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και μπορούν να προληφθούν. Όπως γνωρίζουμε, οι ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις από κοινού. Υπό την Εσθονική Προεδρία θα συνεχίσουμε προωθώντας την ατζέντα υγείας με βάση δύο προτεραιότητες την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ, του ινοπνεύματος, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και την ψηφιακή καινοτομία στην υγεία. Η επιβλαβής χρήση του ινοπνεύματος έχει μεγάλη σημασία για την κοινωνία, δημιουργεί έγκλημα, βία, χαμηλή εργασία και προβλήματα με τα παιδιά και τις οικογένειες. Από όσο γνωρίζουμε υπάρχουν 200 ασθένειες που σχετίζονται με τον αλκοολισμό και το κόστος που αναλαμβάνει η κοινωνία είναι, ανέρχεται στα 272 ε, δις ευρώ. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν ε, το, τον χρόνιο αλκοολισμό και τον ε, διακεκομένο Έχουμε όμως ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι αρχικά προβλεπόταν τα τελευταία 15 χρόνια δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα μόνο σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις διασυνοριακές πτυχές και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν την υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησε για μια ολιστική προσέγγιση της αντιμετώπισης του αλκοολισμού στο ψήφισμα του Απριλίου 2015. Εδώ θα ήθελα να σταθώ στη διαφήμιση του ινοπνεύματος από τα ψηφιακά μέσα, το οποίο αποτελεί δέλεαρ για τους νέους ανθρώπους. Ενώ οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μία νομοθεσία για τον τομέα αυτό, δεν υπάρχει ολιστική προσέγγιση και επειδή υπάρχει και η ψηφιακή αγορά μειώνει το εύρος των κανονισμών των εθνικών νομοθεσιών και επηρεάζει τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Το γεγονός ότι τα αλκοολούχα ποτά αποκλείονται και εξαιρούνται από τις ε, απαιτήσει ε, σήμανσης δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Ο καταναλωτής πρέπει να πληροφορείται σε σχέση με τα συστατικά καθώς και τη θρεπτική αξία των προϊόντων αυτών. Στην εσωτερική αγορά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί από μία χώρα μεμονωμένα. Υπάρχει και η πρόβλεψη της αυτορύθμισης από την Κομισιόν και τη βιομηχανία, αλλά ξέρουμε ότι η αυτορύθμιση είναι δικαιολογία για να μην κάνουμε τίποτα. Και δυστυχώς παρατείναμε αυτή τη διαδικασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά θα πρέπει να προασπίσουμε και τις αξίες της αγοράς και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να βρούμε κοινέ λύσεις. Εάν υπάρχει κανονισμός και κανονισμοί ε, για την προστασία των καταναλωτών στον τομέα του καπνού, καλλιντικών και ούτω καθεξής. Γιατί να μην ισχύει κάτι τέτοιο και για τα προϊόντα εινοπνεύματος και όπως ισχύει σε όλους τους άλλους τομείς. Και γι' αυτό έχουμε να κάνουμε με ένα διασυνοριακό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Την επόμενη εβδομάδα στο Ταλίν, 20 με 21 Ιουλίου, θα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας και θα ασχοληθούμε και με τις επιβλαβείς συνέπειες του Ινοπνεύματος στις 30 και 31 Οκτωβρίου στο Ταλίν. Στη συνέχεια στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Δεκεμβρίου θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα ολιστικά. Σε σχέση με την ψηφιακή Ευρώπη και την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων, αυτό είναι ένα θέμα ε, οριζοντίων προτεραιοτήτων της Προεδρίας και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της ε, γύρανσης του πληθυσμού και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει επαρκής καινοτομία. Θεωρούμε ότι πρέπει να προωθήσουμε τους στόχους υγείας έτσι ώστε και τα εθνικά συστήματα υγείας να είναι πιο ανθεκτικά και διαφανή. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η πρόσβαση στην πληροφορία για να μπορεί κανείς να διαχειριστεί την υγεία του και επιγραμμικά. Και αυτό αφορά ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες. Γι' αυτό και τονίσαμε το θέμα της πρόσβασης και ελέγχου στοιχείων υγείας επιγραμμικά. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει και συνένεση για να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία για την έρευνα. Χρειαζόμαστε διαλειτουργικά συστήματα υγείας έτσι ώστε να υπάρχει συνδεσιμότητα και καλύτερη διάδραση και στον τομέα της αντιμετώπισης υγείας. Θα πρέπει να είμαστε πιο ευφυείς ως προς τον τρόπο χρησιμοποίησης των δεδομένων ιδιαίτερα σε ένα κλινικό περιβάλλον, αλλά και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν τις ασθένειες ε, που τους πλήττουν. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε ατομικά και συλλογικά ευεργετήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε σωστές διαγνώσεις μέσα στα πλαίσια της ιδιωτικότητας των πολιτών και των ευρωπαϊκών αξιών. Επίσης, μέσα στα πλαίσια της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να προωθήσουμε καινοτόμες λύσεις οι οποίες να προβάλλουν συγκεκριμένα ανοιχτά πρότυπα. Επίσης, η ενδιάμεση αναθεώρηση της Κομισιόν μίλησε για τον, για τον μετασχηματισμό αυτού του πλαισίου της ενιαίας αγοράς, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Τον Ιούλιο στο Συμβούλιο Υπουργών θα συζητήσουμε για τον αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των στοιχείων online από τους ίδιους τους πολίτες. Η διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την υγεία στην ε, κοινωνία, στην ψηφιακή κοινωνία, θα λάβει χώρα στο Ταλίν στις 16 με 18 Οκτωβρίου, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τις ε, γενικότερες συζητήσεις για να μπορέσουμε να διαδράσουμε σε αυτή την αγορά το να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων και να ορίσουμε τα πλαίσια υγείας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που προβλέπονται για το Δεκέμβριο, για το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Σε σχέση τώρα με τα, ε, τα προϊόντα που αφορούν το γενικότερο πακέτο ιατρικών προϊόντων, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, πιστεύω, μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Ε, τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαλτέζικη Προεδρία και τις Προεδρίες της Ολλανδίας και της Σλοβακίας για την εξαιρετική τους εργασία. Θα συνεχίζουμε και να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της ε, αντίστασης κατά των μικροβίων και την αντιμετώπιση της φυματίωσης και HIV. Σε σχέση με την ε, αντιμικροβιακή αντίσταση θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μία ε, ολιστική προσέγγιση του AMR και γι' αυτό θα το προωθήσουμε και στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας και στο Συμβούλιο Αγκριφή τον Ιούλιο. Στι 23 Νοεμβρίου προβλέπεται το ε, τελικό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Οι μολυσματικές ασθένειες όπως το HIV, η φυματίωση και η πατήτηδα γάμα ε, μπορούν να επιδράσουν πολύ την κατάσταση υγείας στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διεθνή δεδομένα έτσι ώστε μέσα στα εθνικά συστήματα υγείας να αντιμετωπιστούν το AIDS καθώς και η φυματίωση και να δοθούν βιώσιμες λύσεις. Προβλέπεται μία συνάντηση στις 12 και 13 Δεκεμβρίου για το θέμα μέσα στα πλαίσια και της ε, δήλωσης ε, της Μάλτας για το AIDS HIV και τα συμπεράσματα του ΠΟΗ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αφοσίωσή σας και για την εργασία σας που έχει μεγάλη σημασία για την προάσπιση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την εισήγησή σας και τις ε, προτεραιότητες που παρουσιάσατε πολύ σαφώς. Δίνω το λέω στους συναδέλφους. Καταρχάς θα ακούσουμε τους συντονιστές από τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Λίσε από το ΕΛΚ πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για την ε, εισαγωγική αυτή παρουσίαση. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της παρουσίασης του συναδέλφου σας σήμερα το πρωί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και της δικής σας παρουσίασης. Θα πρέπει από κοινού να φροντίσουμε ε, να αλλάξουν τα πράγματα. Ο συνάδελφός σας το πρωί μίλησε για την κλιματική αλλαγή, για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε στην ημερήσια διάταξη για το περιβάλλον. Εκτός από τα κτηνιατρικά φάρμακα και σας παρακαλώ επ' αυτού το συντομότερο δυνατόν να θέσετε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο διότι χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και θα πρέπει και οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου να ληφθούν υπόψη και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε με τον τριμερή διάλογο. Αλλά αυτό ε, είναι το μόνο το οποίο ε, μπορεί να έχει κάποια ε, πρόοδο από νομοθετική πλευρά. Και ο Ζων Κλοντ Ιούνκερ είχε πει πριν από ε, λίγε μέρε ότι ε, δεν μπορεί να μην υπάρχει νομοθετική πρόταση στον τομέα της υγείας από τότε που υπάρχει η νέα επιτροπή Juncker και Timmermans και αν ρωτήσετε έναν νέο τι θεωρεί πιο σημαντικό, την υγεία θα αναφέρει μεταξύ των πρώτων. Και αυτό το αποδεικνύουν και στις φυγομετρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε αρμοδιότητες σε όλους τους τομείς, αλλά υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, ούτω ώστε να μην δίνουμε την εντύπωση ότι θέλουμε απλώς ε, να, υποχρεώνουμε τους πολίτες ε, ε, να πιούν ή να φάνε αυτό το οποίο θέλουμε. Ο γιος μου με ρώτησε τις προάλλες γιατί γράφει παντού τον αριθμό των θερμίδων και δεν το γράφει πάνω στο μπουκάλι της μπύρας ή σε άλλα αλκοολούχα ποτά. Να, ένα τομέα που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε νομοθεσία. Όπως και στην αντοχή στα αντιμικροβιακά, χρειάζεται ένα πλήρες νομοθετικό πακέτο ούτως ώστε και στο φύλλο χρήσης ε, προς τον ασθενή να υπάρχουν ε, επαρκείς πληροφορίες. Στον τομέα της υγείας μιλάμε πολύ, αλλά τα έργα δεν συνοδεύουν τα λόγια μας ε, και το θέμα της ψηφιακής υγείας είναι ένα από αυτά που αναφέρατε και ελπίζω ότι θα γίνει κάτι ώστε να λειτουργεί καλύτερα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νταλή εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως εκπρόσωπος ε, της Προεδρίας του Συμβουλίου. Χαίρομαι που αναφέρατε το θέμα ε, της επιβλαβούς χρήσεως του αλκοόλ και το θέμα της ηλεκτρονικής καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Όλους μας ενδιαφέρει η δημόσια υγεία και υπάρχουν τομείς όπου μαζί σας μπορούμε να κάνουμε σημαντική πρόοδο. Θα ήθελα καταρχήν να μιλήσω για τη στρατηγική σχετικά με το αλκοόλ και τις αρνητικές επιπτώσεις του αλκοόλ που ξέρω ότι σας είναι ιδιαίτερα προσφυλές θέμα. Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια νέα στρατηγική για το αλκοόλ σχετικά γρήγορα και πιστεύετε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για σωστή επισήμανση των αλκοολούχων ποτών. Και ενώ όλα τα αλκοολούχα ποτά, αλκοολούχα, μπύρες, κρασί κλπ. Αναφέρετε επίσης και την αντοχή στα αντιμικροβιακά. Είπατε ότι θα συνεχίσετε τη συζήτηση. και η Επιτροπή έχει προτείνει ένα σχέδιο δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντοχή στα αντιμικροβιακά. Και θα ήθελα να μας πείτε τι δράση σκοπεύει να λάβει η Προεδρία σας. Πώς σκοπεύετε να προωθήσετε αυτό το θέμα. Ώστε να έχουμε πραγματικά ε, κάποια σημαντική πρόοδο. Όσον αφορά την ψηφιακή υγεία, Μιλήσατε για συντονισμό και συνεργασία για την ηλεκτρονική υγεία. Επίσης αναφέρατε καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στα στοιχεία της υγείας τους, διασφαλίζοντας το ιδιωτικό απόρριτο. Όταν έχουμε και θέματα προστασίας δεδομένων, προκύπτουν ζητήματα τα οποία δεν είναι εύκολα. Πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ανταλή. Ο κύριος Πίρκερ, εκ μέρους της ομάδας ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Η πολιτική μας ομάδα χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες, ε, τις ε, προτεραιότητες τις οποίες θέσατε ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας. Ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές ότι θεωρούμε σημαντικό το θέμα αυτό. Έχουν ληφθεί κάποια αρχικά έχουν γίνει κάποια αρχικά βήματα, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει πολύ. Αναφέρεται και το αλκοόλ και την κατανάλωση αλκοόλ. Αποτελεί ένα προϊόν γεμάτο τοξίνες και ξέρω ότι καταναλώνεται από τους πολίτες και η άμετρη κατανάλωση αλκοόλ έχει επιπτώσεις ε, και στην υγεία και στην κοινωνία. Χαίρομαι ιδιαίτερο λοιπόν που αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας σας, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχω και δύο ερωτήσεις. Πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτά που έχει ξεκινήσει η Προεδρία της Μάλτας ασχολήθηκαν αρκετά με τα θέματα των φαρμάκων. Υπάρχουν, ε, πολλές, ε, πολλοί, υπάρχουν πολλοί δημοσιονομικοί περιορισμοί και πολύ συχνά υπάρχουν ε, παραποιημένα φάρμακα που έχουν επιπτώσει στην υγεία μας. Όσον αφορά λοιπόν τις προτεραιότητές σας, μπορείτε να μας πείτε αν θα λάβετε μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν την αγωγή των ασθενών με φάρμακα τα οποία είναι διοομοειδή. Ακόμη όσον αφορά την καταγραφή ιστών και αίματος. Ε, έχετε κάτι στις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Για τη σύνθεση του αίματος είχαμε μια αρχική οδηγία, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές σε θέματα ασφάλειας. Έχουμε πολύ καλύτερη ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Έχουμε και αυτόματες δοκιμές, έχουμε περισσότερα δεδομένα και είναι πιο εύκολο για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες της υγείας. Η ερώτησή μου είναι κατά πόσο πρόκειται η Αστυνομική Προεδρία να παρακολουθήσει την κατάσταση αυτή, αν θα ξεκινήσετε ένα διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να εξασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας όσον αφορά το αίμα, τους ιστούς και τα κύτταρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χέρκα. Κυρία Κονέτσνα, από μέρους της ΓΚΟΕ. Αγαπητέ Υπουργέ, μια πολύ επίκαιρη ερώτηση. Συμφωνώ με το πρόγραμμα που παρουσιάσατε. Όλοι συμφωνούμε ότι ανάμεσα σε αρμοδιότητες των Υπουργών Υγείας, εσείς έχετε επιλέξει τα πιο επί... Ε, επίκαιρα θέματα. Παραδείγματο χάρη, μικροβιακή εντοχή. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχει παρουσιαστεί και από τι προηγούμενε προεδρίε. Σα εύχομαι λοιπόν εσεί να καταφέρετε επιτέλου να γίνει κάτι για αυτό το θέμα. Θα ήθελα όμω να θέσω ένα πρόβλημα γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση της υπατήτητας C, της φυματίωσης και του AIDS. Έχουμε 30.000 νέες μολύνσεις, νέα περιστατικά δηλαδή, κάθε χρόνο. 120.000 άνθρωποι πάσχουν από φυματίωση. Και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είμαστε, δεν είμαστε θέση να υποχρεώσουμε την Κομισιόν να κάνει κάτι. Θα σας κάνω έκκληση λοιπόν. Εσείς που έχετε την Προεδρία του Συμβουλίου να μας βοηθήσετε για να ασκήσουμε περισσότερη πίεση στην Κομισιόν. Γιατί η Κομισιόν μας είπε ότι σε λίγο, μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή, θα λάβουμε ένα σχέδιο. Δεν θα είναι καν σχέδιο δράσης. Μπορεί να είναι μια δήλωση είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση ως προς αυτό το θέμα. Το πώς δηλαδή αντιμετωπίζουμε την υγεία των πολιτών μας. Είναι ανεπαρκής η δράση μας. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν εδώ απέτυχε. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε βέβαια. Υιοθετήσαμε ένα πολύ σαφές ψήφισμα. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω εσάς, που είσαστε η Προεδρία να προωθήσετε αυτό το θέμα και να πιέσετε την Κομισιόν γιατί δεν μπορούμε εμείς να τα καταφέρουμε χωρίς την υποστήριξή σας. Ο κύριος Eichhout από τους Πράσινους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ που ήρθατε σήμερα το απόγευμα εδώ. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Πίτερ Λίζε ότι το χαρτοφυλάκιο δεν προκαλεί τόσο την περιέργεια του κόσμου. Βλέπετε, έχετε λιγότερου ευρωβουλευτέ, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντικό. Βέβαια δείχνει ότι οι αρμοδιότητες ε, στον τομέα αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι λίγο πιο προβληματικές εδώ. Αυτό δεν βοηθάει, αλλά ελπίζω για κάποια από αυτά τα θέματα εδώ να συνεργαστούμε καλά. Μία συγκεκριμένη ερώτηση έχω να υποβάλω, όπως ε, είπε και η κυρία Ντάρλη. Η μικροβιακή αντοχή. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Κανονικά τι γίνεται. Η Κομισιόν ετοιμάζει ένα έγγραφο, υποθέτω τον Ιούνιο, αλλά στην επόμενη εβδομάδα έχει μπει στην ατζέντα του Συμβουλίου Γεωργίας και Ελίας. Να ένα πρόβλημα. Αν διαβάσετε την έκθεση της Κομισιόν, εξετάζει κυρίως εναλλακτικέ στην πραγματικότητα. Εναλλακτικέ λύσεις, εναλλακτικά αντιβιωτικά καλύτερα. Αλλά η έρευνα δείχνει και περισσότερο ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην χρήση των φυτοφαρμάκων από τη μία και την χρήση των αντιβιωτικών από την άλλη. Επίσης, κάποια, κάποιοι ερευνητέ λένε ότι η χρήση των ζυζανιοκτώνων όταν εξετάζεται χωριστά, σαν χωριστό θέμα, μπορεί να υποτιμά την αύξηση της μικροβιακής αντοχής που υπάρχει. Όταν μπαίνει στην ατζέντα του Υπουργείου, ε, των Υπουργών Γεωργίας και Αλίας, πραγματικά φαίνεται εμφανώς το πρόβλημα που έχουμε. Εσείς ως Υπουργός Υγείας, Καλό θα ήταν να μα πείτε συγκεκριμένα πώ αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ούτω ώστε αυτά τα θέματα να αντιμετωπιστούν μαζί. Να μην τα αφήσουμε μόνο ω θέμα των Υπουργών Γεωργίας, να το δούμε και από τη σκοπιά των Υπουργών υγεία. Ευχαριστώ κύριε Ντορμανό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τον αλκοολισμό, ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα της Προεδρίας σας. Η κατανάλωση, η μαζική του αλκοόλ, είναι υπεύθυνη για πάνω από το 7% ασθενειών και θανάτων. Δηλαδή 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Κάτι που σημαίνει μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ε, καταρχάς πουλάμε το αλκοόλ πολύ φθηνά, το έχουμε εντοπίσει εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γίνεται και διασυνοριακή πώληση αλκοολούχων ποτών στο ίντερνετ. Πρώτη ερώτηση. Σκοπεύετε να προωθήσετε μέτρα κατά αυτών των δύο φαινομένων που προωθούν τον αλκοολισμό. Επίσης, κατ' επανάληψη, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο είχαν διστάμενες απόψεις για το θέμα των γάμματα φόμικρων. Πρόσφατα ένα ψήφισμα προωθήθηκε για να αντιταχθούμε στο σχέδιο της Κομισιόν να θέσει στην ε, εμπορία προϊόντα με γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο. Εμείς ζητάμε τροποποίηση της αδειοδότησης των γαματαφόμικρων γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα και ελλείψεις και τα έχουν καταγγείλει οι ερευνητές. Δεύτερη ερώτησή μου λοιπόν είναι, σκοπεύετε να στηρίξετε τη θέση του Κοινοβουλίου για να εμποδίσετε την Κομισιόν να περάσει καταναγκαστικά ε, κάτω από την πόρτα, έτσι, από το παραθυράκι, το θέμα των γαματαφόμικρων. Κλείνει εδώ ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Υπουργέ, εάν είσαστε έτοιμος, μπορείτε να απαντήσετε τώρα. Αυτέ ήταν οι ερωτήσει των συντονιστών που ακούσατε. Σα ακούμε. Ευχαριστώ για τι παρατηρήσει και τι ερωτήσει. Όπω είπε ο κ. Πίτερ Λίζε καταρχάς, πολύ σωστά διαπιστώνει ο κ. Λίζε ότι Γίνονται πολύ λίγα πράγματα στον τομέα της υγείας. Πολλά προβλήματα όμως υπάρχουν. Ίσως μερικές φορές ε, οι αρμοδιότητες ε, είναι σε διάφορα επίπεδα, από διάφορα, διάφορους φορείς ε, που χρονοτριβούν κτλ. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και τι παίζει με τα κράτη-μέλη. Μερικές φορές το πρόβλημα ναι είναι κοινό, αλλά βλέπετε ότι οι λύσεις δεν είναι εύκολες να βρεθούν σε κοινό επίπεδο. Παραδείγματο χάρη πολιτική για το ενόπνευμα είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Η... Μία συνάδελφο ρώτησε, η ε, κυρία Ντάλη, ε, να, να της πω πόσο εμπιστοσύνη έχω και πόση πρόοδο μπορεί να σημειωθεί. Ε, εμείς ζητάμε ε, στρατηγική από την Κομισιόν, πολλές προεδρίες δηλαδή το ζήτησαν να κάνει κάτι η Κομισιόν, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Ε, ενώ το αλκοόλ κάνει βλάβη στην ε, Ευρώπη και παρόλα αυτά πολλά κρατήμελη δεν υποστηρίζουν κάποια δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι σαφής λόγος γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά γενικά κάτι πρέπει να κάνει παραπάνω η Ευρώπη στο μέλλον από αυτά που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Μην ξεχνάτε ότι τα θέμα τη υγεία είναι τμήμα του κοινωνικού πυλώνα. Ίσως μέσα σε μια πρόταση αυτό απεικονίζεται, αλλά είναι μια σημαντική πρόταση και θα γίνουν και μελλοντικέ συζητήσεις για αυτό το θέμα. Να απαντήσω τώρα σε κάποιες από τις πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και την ψηφιακή υγεία. Φυσικά, Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται κατά της καινοτομία στον τομέα της υγείας. Δηλαδή ότι είναι ευαίσθητα δεδομένα και οι κυβερνήσεις δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσουν στεναρά συστήματα τόσο ότι τα χρησιμοποιούνται σωστά χωρίς ε, καταχρήσεις και προβλήματα. Αυτή είναι μια αντίρρηση όχι κατά του συστήματος τόσο πολύ όσο δείχνει την ανάγκη για να εφεύρουμε τέτοια στεναρά συστήματα προστασία των δεδομένων, τόσο ώστε ο κόσμος να μπορεί να ελέγχει τα δικά του δεδομένα και να μπορεί να τα χρησιμοποιεί και προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και προς όφελός του. οι νομοθέτε ε, υιοθέτησαν σημαντικές νομοθετικές πράξεις πρόσφατα για αυτό το τομέα που κατά την άποψή μας δημιουργεί το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων. Τώρα χρειάζεται να εστιάσουμε στην γρήγορη εφαρμογή του, κανονισμού, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων, ε, την οδηγία για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων. Θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε εδώ και βεβαίως να εμβαθύνουμε την ε, συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για να έχουμε συγκλίνοντα πρότυπα για την ε, κυκλοφορία των δεδομένων. ούτως ώστε να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια διασυνοριακά. Ω προς τη μικροβιακή αντίσταση, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα όχι μόνο από πλευράς υγείας, αλλά και από πλευράς γεωργίας. Και έχει μεγάλη σημασία να προβάλλουμε μια στρατηγική υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει και ένα πρόγραμμα δράσης. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί και στο Υπουργείο Γεωργίας, αλλά και οι Υπουργοί Υγείας θα συζητήσουν το ζήτημα τον Ιούλιο. Η Κομισιόν θα μας υποβάλει ένα πρόγραμμα δράσης την επόμενη εβδομάδα. Όπως σας είπα, προβλέπουμε μία συνάντηση στις 23 Νοεμβρίου του 2017 εδώ στις Βρυξέλλες σε σχέση με θέματα μικροβιακής αντοχής και σε σχέση με τα ε, κτηνιατρικά προϊόντα θα πρέπει να γίνει επιπρόσθετη εργασία στο Συμβούλιο και θα πρέπει να επιταχύνουμε αυτή τη συζήτηση, αυτές τις συζητήσεις, έτσι ώστε στο τέλος της Προεδρίας να έχουμε μια εντολή ως βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και φυσικά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ω ε, ως προς ζητήματα που έχει θίξει το Κοινοβούλιο. Σε σχέση με το HIV, βεβαίω η Εσθονία επειδή έχει τα υψηλότερα ποσοστά σε επίπεδο ενηλίκων στην Ευρώπη, ε, γνωρίζει ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα και εθνικά, ιδιαίτερα για τις χώρες που δεν πέρασαν από τη φάση του δωρητή στην ε, ε, εγγραφή και εφαρμογή του συστήματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και ως διασυνοριακή απειλή. Ξέρουμε ότι η Μαλτέζικη Προεδρία ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα και θα συνεχίσουμε αυτή την εργασία. Και αυτό θα το θίξω και με τον αρμόδιο επίτροπο. Και θα ε, οργανώσουμε ένα σεμινάριο υψηλού επίπεδου στο Ταλίν για να συζητήσουμε αυτό το θέμα της ε, αντιμετώπισης δηλαδή του HIV. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα προχωρούμε στο δεύτερο γύρο με τα μέλη. Ο κύριος Πέτερλε είναι ο πρώτος ομιλητής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να σας συγχαρώ, να συγχαρώ την ανάληψη της πρώτης ε, Εστονικής Προεδρίας. Στην εισήγησή σας ε, υπογραμμίσατε πολλά ζητήματα τα οποία με βρήκαν σύμφωνο, δηλαδή καταρχήν το ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και τι χρησιμοποιούν. Και γι' αυτό ε, τονίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και την ηλεκτρονική ε, υγεία. υγεία. Και να δούμε τι μπορεί να γίνει χωρίς να αλλάξουν οι συνθήκες. Η ηλεκτρονική υγεία μας ανοίγει νέους ε, ορίζοντες που δεν μπορούσαμε καν να έχουμε υποψιαστεί. Μιλάμε για μια ευρύτερη συμμαχία στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας. Και επίσης ε, χαίρομαι για τη δέσμευσή σας ε, ως προς την προστασία των εργαζομένων για τις, ε, έναντι των καρκινογόνων ουσιών. Τον προηγούμενο μήνα με εμπειρογνώμονες προετοιμάσαμε μία εκδήλωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ευρύτερη γνώση, γιατί δεν πρέπει να, να ξεχνάμε ότι 20 εκατομμύρια ε, εκτίθενται σε αυτή τη μορφή καρκίνου και έχουμε και 100.000 θανάτους εξαιτίας αυτής της νεοπλασίας. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε ε, ανώτατα όρια για τους μεταξε, μεταλλαξιογόνους και καρκινογόνους παράγοντες και ουσίες με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τη δυνατότητα μέτρησης έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες. Επίσης, θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς θα κάνει η Εσθονική Προεδρία σε σχέση με τις προκλήσεις που μόλις προανέφερα ο κύριος Παρνιό. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, κύριε Υπουργέ, και για τις πρώτες σας απαντήσεις. Έφεξε ένα ζήτημα το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την προστασία των Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών που θα εντάξετε στην εξαμηνία σας ατζέντα. Πρόκειται για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν κριτήρια για την αναγνώριση αυτών των διαταρακτών και λυπάμαι γιατί μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων 21 κράτη-μέλη, εκ των οποίων και η Γαλλία, προβάλλουν κριτήρια τα οποία τάσσονται υπέρ της βιομηχανίας και όχι τόσο υπέρ των πολιτών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να ορίσουμε πολύ ε, καλύτερα έναν ενδοκρινικό διαταράκτη θέτοντας χαμηλότερα και όχι τόσο υψηλά ε, όρια. Υπάρχουν η πληθώρα εξαιρέσεων και το Βερολίνο ζήτησε εξαιρέσεις σε σχέση με τα παρασιτοκτόνα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν, να οδηγήσουν σε αυτούς τους ενδοκρινικούς διαταράκτες στον άνθρωπο και στα ζώα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις μήνες για να λάβει θέση σε αυτή την ε, αρχική πρόταση της Κομισιόν. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε κύριε Υπουργέ κατά πόσο είσαστε ικανοποιημένος από αυτή την πρόταση και αν όχι πώς θα ξαναθέσετε την υγεία στο επίκεντρο των μελημάτων σας με βάση την αρχή της πρόληψης. Ευχαριστούμε πολύ. Φαρία. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Το πρωί είχαμε τη χαρά να καλωσορίσουμε τον συναδελφό σας, τον κύριο Κίσσερ, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όπως γνωρίζετε, ο κίνδυνος ε, της μικροβιακής αντοχής ε, για τη δημόσια υγεία και για και οι οικονομικές συνέπειες ε, που θα είναι επίπτωση αυτού αυξάνεται συνεχώς. Πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα για νέα αποτελεσματικά αντιβιωτικά και θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ασθενείς όλων των ηλικιών θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες οι επενδύσεις ε, που συνεχίζονται στην έρευνα και στην ανάπτυξη για νέα αντιβιωτικά θα πρέπει να ε, ε, χρησιμοποιούν ήδη τα υφιστάμενα στοιχεία και τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα έρευνας. Ως Υπουργό Υγεία και υπεύθυνο της Προεδρίας του Συμβουλίου, τι μέτρα θα λάβετε για να αντιμετωπίσετε την αντοχή στα αντιμικροβιακά και ποιες είναι οι προτεραιότητες της Εσθονίας για τα γενώσιμα και τα βιομοειδή. Από το 2013 υπάρχει ε, μια στασιμότητα στα θέματα της στρατηγικής για το αλκοόλ. Τι θα κάνετε, θα συνεχίσετε μαζί με την Επιτροπή να καθυστερείτε ή θα καταβάλλετε προσπάθειες για να πιέσετε την Επιτροπή να λάβει ενεργό δράση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φαρία. Η κυρία Καβεσόν Ρουίς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Νομίζω ότι γίνεται λόγο ε, πρωτίστω για το... Αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το ινοπνεύμα αλλά και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Μιλήσατε και για το νέο πρόγραμμα δράσης κατά της ε, μικροβιακής αντοχής και το e-health. Ως προς τη μικροβιακή αντοχή θα, θέλουμε, θα θέλαμε να προωθήσουμε και τα εθνικά πρόγραμματα. Το πρώτο θέμα είναι Πώ ε, θα είναι ένας δεσμευτικός στόχος ή υποχρεωτικά εθνικά σχέδια, γιατί δεν ξέρουμε καν σε ορισμένα κράτη-μέλη πώς κάνουν χρήση αντιβιωτικών πριν, ε, πριν γίνει ενδελεχής έρευνα. Πώς μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε τα εθνικά προγράμματα χρήσης των ε, αντιβιωτικών και τι συντονισμός γίνεται. Μιλάμε επίσης και για ε, σπάνιες ασθένειες και την αντιμετώπιση τους και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συντονίσουμε τις δημόσιες προσπάθειες σε σχέση με το, την ηλεκτρονική υγεία φτάνουμε σε ριζοσπαστικά στοιχεία αλλά θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και η διακυβέρνηση των δεδομένων. Μιλάμε για το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων, αλλά υπάρχει και το δικαίωμα εκμετάλλευσης των δεδομένων. Ποιοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, να τα ελέγξουν, να τα χρησιμοποιήσουν μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και ποιο είναι το ευεργέτημα για τους ασθενείς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ε, δύο ε, συστήματα υγείας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το να μιλάμε για διακυβέρνηση δεδομένων έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής ε, ατζέντας. Περιμένουμε επίσης και τη μελέτη αντικτύπου έτσι ώστε να προωθήσουμε τα δεδομένα που υπάρχουν και να δούμε ποια είναι και τα ε, νέα ιατρικά δεδομένα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στα πλαίσια ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε την αξιολόγηση των φαρμάκων μέσα στα πλαίσια της ε, υγείας. Ευχαριστούμε πολύ. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich danke auch erstmal sehr herzlich, ähm, Herr Minister, dass Sie Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, Υπουργό που δίνει το χρόνο και που έρχεται εδώ να συζητήσει μαζί μας. Μίλησε και ο Πέτερ Λίζα για αυτό το σημείο. Και όλοι οι συνάδελφοι, νομίζω, ενδιαφέρονται και ανέφεραν αυτό το θέμα, την αντοχή στα αντιμικροβιακά, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα. Συνεχίζοντας σε σχέση με αυτό που ανέφερε ο Πέτερ Λίζε, Φαίνεται ότι τα κτηνιατρικά φάρμακα είναι μακριά από την ανθρώπινη υγεία, κάθε άλλο όμως όλα σχετίζονται. Και είναι πολύ σημαντικό και το θέμα των κατάλοιπων ε, αντιβιωτικών. Επίσης πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και με τα online φάρμακα μέσω διαδικτύου. Είναι θέματα που απασχολούν και εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2016 συζητήσαμε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν η Εσθονική Προεδρία μπορεί να συνεισφέρει, θα είναι για μας ιδιαίτερα θετικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Φουντούλης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα εντάξετε στην ατζέντα σας το θέμα του αλκοόλ. Ε, ο αλκοολισμός τίνει να γίνει μια μάστιγα στην εποχή μας και ειδικά στους νέους όπως είναι τα ναρκωτικά, ε, έτσι έχουν εξελιχθεί και ο αλκοολισμός. Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση. Όπως τα πακέτα από τα τσιγάρα έχουν μπει κάποια μπάνερα από κάτω και προειδοποιούν ότι το τσιγάρο σκοτώνει, ε, αυξάνει την ε, υπογεννητικότητα, δημιουργεί ασθένειες. Γιατί να μην υποχρεώσουμε και τις εταιρείε επάνω στα, μπουκάλια να γράφουν ότι ο αλκοολισμός είναι εθισμός ότι όταν οδηγείς υπό την επίρρη αλκοόλ θα σκοτωθείς ή εσύ ή κάποιοι άλλοι. Αυξάνει την, τη βία και ιδιαίτερα την ενδοοικογενειακή βία. Λοιπόν, ξέρω ότι τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ μεγάλα και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ε, οι εταιρείε θα αντιδράσουν σίγουρα. Αλλά όταν βομβαρδιζόμαστε στην τηλεόραση από διαφημίσεις που διαφημίζουν το αλκοόλ και δείχνουν στην νεολαία ότι η ζωή είναι ένα πάρτι θα πρέπει να μπει ένα φρένο. Δεν αρκεί ένα μικρό μπανεράκι ότι καταναλώνω υπεύθυνα. Πρέπει να γίνει μια ενημέρωση. Και όσον αφορά το, το HIV και το AIDS, τα οποία κρούσματα έχουν αυξηθεί, ε, συγκεκριμένα στη χώρα μου την Ελλάδα, έχουν επανεμφανιστεί ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί προπολών ετών, όπως είναι η φυματίωση. Μήπω θα πρέπει να δοθεί μια έμφαση σε όλους αυτούς τους μετανάστες που έρχονται προς την Ευρώπη να ελέγχονται, γιατί δυστυχώς έχουν έρθει πάρα πολλές ασθένειες, σας είπα όπως είναι η φυματίωση, και είναι σε έξαρση και νοσούν και άνθρωποι που ασχολούνται εκεί με την προστασία τους και την περίθαλψή τους. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. If uh, any uh, of the colleagues present today would like... Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Αν όχι, Υπουργέ, έχετε ένα πακέτο ερωτήσεων να απαντήσετε. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Καταρχήν, για το αλκοόλ. Και βέβαια το Συμβούλιο θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στην Επιτροπή να αναλαμβάνει ενεργοδράση. Και όπως σας είπα, είναι ένα από τα θέματα όπου μεταξύ των κρατών μελών διαφέρουν οι απόψεις για να, πει, για να πω στο δυνατόν να περιγράψω στο δυνατόν πιο ήπια την κατάσταση. Υπάρχει η οδηγία για τα προϊόντα καπνού και γνωρίζετε πολύ καλά ότι πριν από 20 χρόνια δεν θα διανοεί το κανείς ότι θα είχαμε μια τέτοια οδηγία για προϊόντα καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της τεράστιας πίεσης από τον κλάδο. Αλλά μετά από πολλές μάχες κέρδισε η δημόσια υγεία. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και με το αλκοόλ. Αλλά οι μάχες μόλις έχουν ξεκινήσει. Είναι σημαντικό τα σημαντικά αυτά θέματα να τα διατηρήσουμε στο θεματολόγιό μας και αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Όσον αφορά τη χρήση δεδομένων, θέσατε το θέμα της πρόσβασης στα δεδομένα και της ακαιρεότητας των δεδομένων. Και βέβαια, τα, επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά της ηλεκτρονικής υγείας είναι ότι είναι ευαίσθητα δεδομένα για την υγεία και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα στεναρό πλαίσιο για την ασφάλεια των δεδομένων. Διαφέρει η παράδοση που ακολουθείται σε κάθε κράτος μέλος και χρειάζεται και κάποια προφύλαξη στη σχέση σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων υγείας, αλλά όλα αυτά θα αποτελέσουν το κλειδί για ένα αποτελεσματικό σύστημα. Στην Εστονία, παραδείγματο χάρη, μόνο οι γιατροί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ηλεκτρονικά δεδομένα για την υγεία. Χρειάζονται δηλαδή πολύ αυστηροί περιορισμοί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα που θα το εμπιστεύονται οι ασθενεί. Για του ενδοκρινικού διαταράκτε, Αρχές Ιουλίου, στη μόνιμη Επιτροπή Ζωοτροφών, ψήφισαν τα κράτη-μέλη υπέρ του κανονισμού και όταν ε, ε, η Επιτροπή στείλει τα αντίστοιχα κείμενα θα υπάρχει και το δικαίωμα ελέγχου και θα μπορέσετε να εξετάσετε τα κείμενα αυτά. Για την πρόσβαση στα φάρμακα Ξέρετε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά και αμφιλεγόμενο. Έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη για την εκούσια συνεργασία και πιθανές ε, δράσεις αφορούν ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών για θέματα τιμολόγησης και αποζημίωσης και η Επιτροπή εξετάζει πιθανά κίνητρα προς τη φαρμακευτική βιομηχανία και εξετάζει και θέματα διαθεσιμότητας φαρμάκων. Η Εστονική Προεδρία θα εξετάσει το θέμα της πρόσβασης στα φάρμακα σε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου για τη φαρμακευτική πολιτική, όπου θα εστιάσουμε σε θέματα συνεργασίας. Το θέμα της μικροβιακής αντοχής συζητήθηκε πολλές φορές. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Χαίρομαι που η Επιτροπή έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης και αυτό είναι άλλο ένα θέμα όπου απαιτείται δράση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι σοβαρό το πρόβλημα το ότι, του ότι δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα σε πολλές χώρες και εδώ μπορεί να μας βοηθήσει η ηλεκτρονική υγεία. οι συνταγέ αντιβιωτικών και για ανθρώπους αλλά και για ακτινιατρικά φάρμακα θα μπορούσαν ε, αυτόματα ε, να καταγράφονται αν είχαμε ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία από τις πρωτοβουλίες για την ψηφιακή υγεία. Όχι μόνο για τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση, αλλά και για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Η ψηφιακή υγεία λοιπόν εδώ θα μας βοηθούσε στην τήρηση στατιστικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας και για άλλα θέματα. Και ελπίζω ότι θα έχουμε επικοδομητική συνεργασία κατά την Προεδρία μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία κατά την Προεδρία σας και προσβλέπουμε και εμείς σε μια πολύ καλή συνεργασία. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η έκθεση της κυρίας Αγιούσο για τον ορισμό παρουσίαση και σήμανση αλκοόλουχων ποτών. Πρόκειται για το σχέδιο γνωμοδότηση και καταρχήν δίνω το λόγο στην κυρία Αγιούσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτός ο κανονισμός, αυτή η πρόταση κανονισμού τροποποιεί τον κανονισμό του 2008 για να τον προσαρμόσει. Πρόκειται για την ομογενοποίηση των προϊόντων αυτών σε σχέση με τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά καθώς και τα τρόφιμα για να προσαρμοστούν στη συνθήκη της Λισαβόνας. Μία ε, αλλαγή είναι το άρθρο 42, παράγραφος 2, για να τονίσουμε το γεγονός ότι πρόκειται για γεωργικά προϊόντα, κάτι το οποίο δέχομαι. Βεβαίως έπρεπε να προσαρμοστεί αυτή η νομοθεσία για να συμβαδίσει με τα νομικά μέσα της συνθήκης της Λισαβόνας. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει όλη η διαδικασία προσαρμογής να λάβει υπόψη τα προνόμια που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει της νομοθεσίας για τη ρύθμιση γι' αυτό Έχω υποβάλει τροπολογίες για κατεξιοδότηση πράξης για να προστατευτούν τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί που προβλέπονται τροποποιήσεις υπό έλεγχο για να συμβαδίσουμε ε, με την περίπτωση που υπάρχουν κατεξιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις. Πρόκειται για ουσιαστικά στοιχεία του κανονισμού και θα πρέπει αυτές οι δεσμεύσεις να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα, μιλάμε για πέντε χρόνια δηλαδή, ε, δυνα... με δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε χρόνια. Πρόκειται για μια ουσιαστική τροποποίηση και πρόκειται για αλλαγές στο κεφάλαιο 3 που διέπουν τις, ε, το γεωγραφικό προσδιορισμό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε συγκεκριμένα καθεστώτα εφαρμογής. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν ιδιάζοντα τομέα. Μιλάμε δηλαδή για τα αλκοολούχα ποτά και έχω υποβάλει τροπολογίες έτσι ώστε ο γεωγραφικός προσδιορισμός με βάση και τις ε, τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να προστατεύεται από τον τρέχοντα κανονισμό, δηλαδή μόλις τεθεί σε εφαρμογή. Μία άλλη από τις τροποποιήσεις είναι η διαγραφή του παραρτήματος 3, εκεί όπου συλλέγουμε όλες τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις με βάση τον κανονισμό 110. Και η πρόταση της Επίτροπης ορίζει ένα ηλεκτρονικό μητρό παρόμοιο με αυτό που ισχύει για την περίπτωση προστασίας της ονομασίας ιδιαίτερα για τα τρόφιμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε και να εξυγχρονίσουμε το σύστημα με αυτό το ηλεκτρονικό μητρό. Υπήρξαν ε, αμφιβολίες, αλλά νομίζω ότι η πρόσβαση γίνεται πιο εύκολη. Επειδή το Μητρό είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία κατάρτισής του και το Κοινοβούλιο. Και εγώ είχα αμφιβολίες σε σχέση με την απαλήφη του παραρτήματος 3, όπως και πολλοί άλλοι, γι' αυτό θα ήθελα και τη δική σας γνώμη. Στο άρθρο 13 της πρότασης αναφέρεται ε, αναφέρονται οι περιορισμοί στο παράρτημα 2 για τα αλκοολούχα που δεν μπορούν, ε, στοιχεία από τα οποία δεν μπορούν να εισαχθούν στη σήμανση. Υπάρχει ένας προγενέστερος κανονισμός, όμως οι τίτλοι δεν γράφονται με πλάγια γράμματα και νομίζω ότι θα πρέπει να συμβαδίζουμε με τον κανονισμό τον οποίο τροποποιούμε. Επίσης έχουν υποβληθεί τροπολογίες στο παράρτημα 2 με στόχο να είναι συνεκτικός αυτός ο κανονισμός με τον ισχύοντα. Τελικά πρόκειται για έναν τεχνικό κανονισμό για να προβεί σε ορισμένες τροποποιήσεις ως προς τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις, εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες, δεν είναι πολλές, αλλά θα ήθελα να μου πούν τη γνώμη τους οι σκιώδεις και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιούσο. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές που είναι παρόντες. Η κυρία Μεριά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστήσω την κυρία Γιούζουα για την έκθεσή της. Έχετε λάβει υπόψη σας πολλές από τις διορθώσεις ε, που έχουμε κάνει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, γι' αυτό. Καταρχήν, θα ήθελα να πω εξ ένα πολύ σημαντικό σημείο όπου πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό για όλους τους συναδέλφους και θα πρέπει και στο μέλλον να το προσέξουμε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως ε, τα μικρά αποστακτήρια μικρών γεωργών ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτή η μικρή ε, παραγωγή θα πρέπει να έχουν δίκαιες ευκαιρίες εμπορίας των προϊόντων τους όταν έρχονται σε ανταγωνισμό με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για να μπορούν να βρουν μια διέξοδο για τα προϊόντα τους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω όμως, θα περιοριστώ σε τρία σημεία μόνο. Όσον αφορά τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις, ε, τα είπατε ήδη κυρία Γιούζο, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Αλλά υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία έχω ε, και εγώ κάποιες τροπολογίες να καταθέσω. είναι θέματα ε, στα οποία έχουμε κατεξουσιοδότηση πράξης. Είναι πολύ τεχνικό αυτό το σχέδιο κανονισμού. Και θα πρέπει να προσαρμοστεί κάπως ε, ο προηγούμενος κανονισμός. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ε, τι θα αφορά πράξεις κατεξουσιοδότηση. το Κοινοβούλιο έχει περιορισμένες εξουσίες όσον αφορά αυτά τα θέματα. Το, η Επιτροπή μπορεί να καταθέσει ένα πακέτο ε, με ε, πολλές κατεξοδότηση πράξεις και εμείς μπορούμε συνολικά να το απορρίψουμε. Ε, ως παράδειγμα να πάρω το άρθρο 5. Μπορούν να τροποποιηθούν τα παραρτήματα με κατεξουσιοδότηση πράξη. Η συγγήτρια θέλει να περιορίζει αυτό το δικαίωμα της Επιτροπής στα πέντε χρόνια. Δεν το θεωρώ επαρκές αυτό. Οι τεχνικοί ορισμοί των αρκολούχων στο παράρτημα 2 αποτελούν σημαντικό τμήμα του κανονισμού. Αποτελούν τον πυρήνα του κανονισμού. Ε, και σύμφωνα με το άρθρο 290 των συνθήκων, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κατεξουδότηση πράξεις. Αυτή η διάταξη, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Και τα τελευταία χρόνια έγιναν πολύ λίγες τροποποίησεις στον κανονισμό ε, για τα αλκοολούχα ποτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια σωστή νομοθετική διαδικασία και είμαι βεβαίω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να τα καταφέρει. Το θέμα της προσθήκης ε, ε, Σακχάρου και η εναρμόνιση των μέτρων επ' αυτού στον κανονισμό αναφέρεται η ε, τροποποίηση της γεύσης με την προσθήκη ε, σακχάρου. Με την προσθήκη σακχάρου ε, μπορούν να διορθώνονται σφάλματα στην διαδικασία απόσταξης, όχι μόνο βελτίωση της γεύσης μπορεί να παρουσιάζεται ως βελτίωση της γεύσης, αλλά δεν είναι πάντοτε αυτό περί του οποίου πρόκειται. Και αυτό με φέρνει και στην ε, τρίτη παρατήρησή μου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με το Συμβούλιο των Υπουργών. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο ζάχαρο περιλαμβάνεται σε ένα, ποτό, σε ένα ποτήρι λικέρ. Έχουν ζητηθεί μέτρα αυτορύθμισης από τους παραγωγούς, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτύχει. διότι είναι διαφορετικά τα συμφέροντα των παραγωγών μπύρας, ίνου ή ίνοπνευματοδών ποτών. Εάν δεν επιτυχεί η αυτορύθμιση θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα και να επιβάλλουμε μια υποχρεωτική επισήμανση. Γιατί σε ένα κοκακόλα να πρέπει να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε σάκχαρο, αλλά όταν η ίδια κοκακόλας προστίθεται στο ρούμι, γιατί δεν αναγράφονται τα συστατικά το ζάχαρο συνεχίζει να υπάρχει και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο καταναλωτής και θα πρέπει να του προσφέρουμε την ενημέρωση αυτή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σαφής ε, επισήμανση με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι τρεις παρατηρήσεις που θεωρώ σημαντικότερες και θα υποβάλω και αντίστοιχες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Γιούσο, για την δουλειά που έκανε. Είμαστε αισιόδοξοι για αυτή την έκθεση, έτσι όπως την είδαμε στην αρχική εκδοχή της. Η εναρμόνιση της ορολογίας μοιάζει να είναι το βασικό θέμα εδώ. Ίσως η ονομασία πώληση. είναι ο όρος που θα έπρεπε να μας απασχολήσει περισσότερο και να, προτιμήσουμε. Γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά ονόματα, εμπορικά ονόματα, ε, κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, όλα είναι πολύ αόριστα και μπορεί να μπερδεύουν πάρα πολύ τον κόσμο και να δημιουργούν πραγματικά χάος Επίσης, αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε, είναι μια διάκριση ανάμεσα στην ορολογία αλκοολούχα ποτά, από τη μία, και ποτά από την άλλη. Έχουμε τροπολογία 5, που αφορά τα αλκοολούχα ποτά, που συμπεριλαμβάνουν και τα ποτά. Θα πρέπει όλα να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Μ' αρέσουν διατάξεις της, υπό την τροπολογία 7 που μιλάει για το να, λυθεί, να λυθούν υπόψη διατάξεις των κρατών μελών. Μ' αρέσει επίσης και η τροπολογία 1 η οποία αναφέρεται στις παραδοσιακές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς, δεν μπορώ να υποστήριξω πλήρως όλες τις περιπτώσεις που γίνεται εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αμφιβάλλω επίσης ε, για πολλές καταξιοδότηση και εκτεταστικέ πράξεις. Τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων, ε, τις αλλαγέ των ορισμών και την προσθήκη ή αφαίρεση ορισμών, αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι που να γίνεται μέσω καταξιοδότηση πράξεων. Θα πρέπει να γίνεται σε πολιτικό επίπεδο. Οι εκτελεστικές πράξεις είναι μάλλον καλύτερη λύση από τις ε, κατεξοδότηση πράξεις. Τροπολογία 16, 18 και 20. Αυτές δηλαδή οι τροπολογίες δεν είναι αρκετά καλές κάτι την απόψή μου. Επίσης, να τονίσω τα εξή. Το μέγιστο επιτρεπόμενο αλκοολούχο αλκοολικό μάλλον περιεχόμενο ή αλκοολικός τίτλος. Αυτό λείπει από το έγγραφο. Για κάποια από τα ποτά όπως η αλκοολικος τιτλο αυτο λειπει απο το εγγραφο για καποια απο τα ποτα οπω η βοτκα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιορισμός. Θα πρέπει να οριστεί αυτό στην τροπολογία 43. Το μέγιστο, ο μέγιστος αλκοολικός τίτλος θα πρέπει να τονιστεί. Και θα πρέπει να έχουμε και περιορισμού σε ό,τι αφορά την ποιότητα τη εθιλικής αλκοόλη. που αντιστοιχεί με τα επίπεδα που αναφέρονται στο παρτιμα 1 1-1. Η ποιότητα του υνοπνεύματος επίσης θα πρέπει να ορίζεται πολύ πιο επακριβώς γιατί οι σχετικές διατάξεις είναι πολύ αόριστες. Προχωρώ τώρα σε άλλα σημεία. Μέγιστο περιεχόμενο σε ζάχαρη, σε κάποια αλκοολούχα ποτά. Δεν είναι αρκετά επακριβές αυτό το στοιχείο. Δεν έχουμε καμία διάταξη που να αφορά το μέγιστο περιεχόμενο σε ζάχαρη για αυτή την κατηγορία ποτών. Επομένως, θα πρέπει να βασιζόμαστε σε, στα όσα αναφέρονται για το, τα αλκοολούχα ποτά με γεύση, όπως ας πούμε τα λικέρ ή η βότκα. Όμως τα γλυκά αλκοολούχα ποτά έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα υπόλοιπα ποτά. Μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουν και διαφορετικές θερμίδες. Σε ό,τι αφορά την προσθήκη ζάχαρης ε, και γλυκαντικών, και εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο ακριβείς. Μιλάμε για τα σημεία 1 έως 4 του παρατήματος. Τα όρια σε ζάχαρη θα πρέπει να αναφέρονται. Παραδείγματος χάρη στο άρθρο 4, σημείο 1. Τα αλκοολούχα ποτά μπορούν να δέχονται περισσότερη δάχαρη, ζάχαρη, ε, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και όρια, γιατί δεν υπάρχουν όρια τώρα στο βαθμό ζάχαρη που προσθέτουμε. Ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και να φτάσουμε σε ενιαία θέση. Γεωγραφικές ενδείξει. Άλλο πρόβλημα αυτό. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που αφορούν τα επιμέρους στατικά. Οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν θα πρέπει να αναφέρονται κατόνομα στον κατάλογο συστατικών λείπει αυτό το στοιχείο από το πάρτιμα, από το, τις τροπολογίες 8 και 9. Επίσης να σας αναφέρω και κάποιους φόβους μου. Ο πρώτος φόβος είναι η διαγραφή του τόπου παρασκευής ή παραγωγής. Ανταυτού έχουμε μια παραπομπή στον τελωνιακό κώδικα. Αυτό όμως είναι προβληματικό, γιατί πολλά αλκοολούχα ποτά ε, τη χάνουν ε, επεξεργασίας πολύ πριν ε, ολοκληρωθεί η Παρασκευή. Και το, ο τελικός τόπος Παρασκευής δεν είναι ο τόπος που πραγματικά παρασκευάστηκε το ποτό αυτό. Παραδείγματο χάρη τα μείγματα ουίσκι, ας πούμε. Το 80% τέτοιων μείγματων είναι σκοτσέζικα. Αλλά το μείγμα, η μίξη, η μίξη μπορεί να γίνει σε ένα άλλο κράτο όχι στη Σκοτία. Ως αποτέλεσμα λοιπόν, ένα τέτοιο ποτό μπορεί να μην θεωρηθεί, ας πούμε, σκοτσέζικο με βάση τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις, έτσι όπως τα προτείνουμε. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολλές περιπλοκές. Πάρα πολλά προβλήματα. Έχω και άλλους φόβους. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 8, παράγραφος 5. Οι μη αλκοολούχες απομιμήχησης και άλλα προϊόντα μπορούν κατόνομα να παραπέμπουν ε, σε ένα είδος αλκοολούχου ποτού. Προσθετικά ή ενισχυτικά γεύσεις. Μπορεί να μπερδέψουν τους καταναλωτές. Μπορεί να θεωρήσουν ότι η βότκα, το ουίσκι και όλες οι ουσίες που αναφέρονται στην ετικέτα να περιλαμβάνονται στο προϊόν. Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν επίσης θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι αυτές οι προτάσεις δεν θα παραπλανούν τους καταναλωτές, ειδικά δεν θα παραπλανούν τα παιδιά. Για να συνοψίσω, το κείμενο είναι αρκετά καλό, αλλά εγώ θα υποβάλω τροποποιήσεις, τροπολογίες συγγνώμη, για όλα αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα. Ευχαριστώ κύριε Πιέκα. Η κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα ευρωπαϊκά αλκοολούχα ποτά έχουν πολύ καλή φήμη σε ολόκληρο τον κόσμο και ε, δικαίως γιατί έχουμε ε, καλά γεωργικά προϊόντα με μακρά παράδοση και γι' αυτό παράγονται τέτοια αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν τέτοιοι μικροί παραγωγοί και στη χώρα μου, στη Γερμανία, αλλά υπάρχουν και σε άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. και αυτό αναγνωρίζεται από το άρθρο 43.2. Είναι σημαντικό να παραμείνει και στο μέλλον σύνδεση του τομέα των αλκοολούχων ποτών με τη γεωργία για να έχουμε ένα ποιοτικό τομέα. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποδώσουμε την απαραίτητη προσοχή για να διατηρήσουμε αυτές τις ε, μικρομεσαίες ε, εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις παραδοσιακές μεθόδους και ήδη έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί σωστά και αποτελεί και βάση για το σύστημα ε, προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να παραμείνουμε στο, ε, στάδιο, στο ένα στάδιο που, που είχαμε μέχρι τώρα ή στα δύο στάδια τα οποία εισάγει η Επιτροπή με την πρότασή της. Αυτό θα το συζητήσουμε κατά τις επόμενες εβδομάδες. Ε, όσον αφορά ε, τα μικρά αποστακτήρια, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο κόστος χωρίς να προσδίδει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. θα πρέπει να προσφέρεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και επίσης ε, σημαντικό είναι για τη διαδικασία της παραγωγής ε, ε, το κατά πόσο θα τηρείται και το δικαίωμα παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας υπενθυμίζω τον κανονισμό για τον ορισμό του αψέντη και εδώ έχουμε κείμενα που αποτελούν ε, και βασικό κανονισμό και παρέμβαση των ε, κατεξοδότηση πράξεων. Ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρώ σημαντικό είναι ότι η χρήση σακάρων μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και σε έλλειψη διαφάνειας για τον καταναλωτή. θα πρέπει από κοινού να προωθήσουμε ποιοτικά πρότυπα. Και θα πρέπει ε, να ε, καταγράφονται αυτά τα αποστακτήρια τα οποία δηλώνουν σαφώς ότι δεν χρησιμοποιούν προστίκη σακχάρεως. Η συγκίτρια στην έκθεσή της έχει διορθώσει αρκετά σφάλματα της Επιτροπής και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά θέματα. Προς τη συνάδελφο Μέλλερ θέλω να πω ότι εδώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια δήλωση ε, όπως αυτή που προτείνατε, γιατί αυτό αφορά περισσότερο ε, τον τομέα των τροφίμων. Διαφορετικά θα έπρεπε να ισχύει για όλα τα αλκοολούχα ποτά. Προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία. Ε, λυπάμαι που θα πρέπει να αποχωρήσω, αλλά και στην Επιτροπή Γεωργίας γίνεται παράλληλα μια συζήτηση με την Εστονική Προεδρία. Θα παρακολουθήσει όμως τη συζήτηση βοηθός μου, οπότε θα μπορέσω να συμμετάσχω στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μιούλε. Η κυρία Μόλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της. Συμφωνώ με τις περισσότερες τροπολογίες που έχει υποβάλει. Πρωταρχικά είναι ένα τεχνικό ζήτημα και μιλάμε για ένα status quo και την απλούστευση και τη διασάφιση των, του κανονισμού. Έχω όμως ορισμένα ζητήματα με την πρόταση της Επιτροπής γιατί υπάρχουν κενά για το μέλλον. Γι' αυτό θα υποβάλω δικές μου τροπολογίες ιδιαίτερα ε, για τα ε, παραχαραγμένα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ με ενδιαφέρει το εμπορικό σήμα. σε σχέση με τις ε, ψεύτικες γεωγραφικές ενδείξεις, κάτι που μας έχει απασχολήσει και στην Ιρλανδία. Επίσης υπάρχει μια πολύ ε, περιοριστική ονομασία ε, των γεωγραφικών ενδείξεων και θα ήθελα στο 8.4β να το ξαναδούμε το ζήτημα. Επίσης, στις ε, ε πράξεις, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ακριβώς με το τι εννοούμε και το ηλεκτρονικό μητρό αποτελεί βεβαίως βελτίωση, αλλά θα ήθελα κάποια μορφή παρατήματος 3 να υπάρχει για τις γεωγραφικές ενδείξεις και όσο αφορά τα αλκοολούχα να μην είναι πολύ επιβαρημένο το σύστημα αλλά υπάρχει μεγαλύτερη νομική προστασία. Ως προς το άρθρο 12 του νέου κανονισμού, νομίζω το ανέφεραν και ορισμένοι σκιώδη σε σχέση με την προέλευση του προϊόντος, νομίζω ότι η εφαρμογή αυτή του άρθρου θα οδηγούσε σε ε, λανθασμένες ενδείξεις σε σχέση με την σήμανση των προϊόντων. Επίσης, σε σχέση με τις ΜΜΕ, αυτός ο κανονισμός δεν πρέπει να τις αφήσει σε μια μειονεκτική θέση, όπως είπαν και άλλοι Εσκιόδης Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής. Έχουμε λοιπόν πολύ καλές βάσεις εργασίας και ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Προσβλέπω σε πολύ καλή συνεργασία. Η κυρία Ντορνανό. Αυτό. Αυτό θα έλεγα, αυτό θα έλεγα, ότι είναι η δική σας σειρά από τους πράσινους. Με συγχωρείτε. Αντικαθιστάτε, κυρία Ετές επί του θέματος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, μιλώ εξ ονόδος του Μπατστάς που είναι σκιώδης από τους Πρασίνους και δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα όπως και όλοι οι άλλοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αγιούσο για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Περιλαμβάνει πολλά καλά στοιχεία αλλά θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε αυτά που θέλουμε εμείς, δηλαδή τα δικαιώματα των καταναλωτών. Μας εκπλήσει το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε σωστές πληροφορίες για τον ε, καταναλωτή ως προς τα αλκοολούχα. Οι δικές μας ζηθοποιίες στη Δανία πάντα μας δίνουν πληροφορίες για το περιεχόμενο της μπύρας. Γιατί είναι τόσο δύσκολο όταν μιλάμε για κρασί και αλκοολούχα. Ζούμε σε μία από τις περιοχές που καταναλώνεται το περισσότερο αλκοόλ. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Εστονός Υπουργός τόνισε ότι χρειαζόμαστε σωστές πληροφορίες για τα ποτά αυτά προς τους καταναλωτές. Μιλάμε για μία Καμινή μη δεσμευτική ε, υπόδειξη και όταν μιλώ με, με εινοπαραγωγούς ε, μου λένε ακριβώς αυτό ότι δεν θέλουν να ενοχληθούν οι εινοπαραγωγοί δεν θέλουν να δώσουν λανθασμένες πληροφορίες πρωτίστως, όμως χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για προσθήκη σακχάρων, για θερμιδική αξία, για ε, αλλεργιογόνες ουσίες και για χρήση εσπεριδοειδών. Χρειαζόμαστε πληροφορίες για όλα αυτά. Στην ε, πρόταση της ε, Επιτροπής Βιομηχανίας θεωρούν ότι τα 30 σεντιλίτρ θα πρέπει να είναι ο γνώμονας, γιατί σε αυτή την περίπτωση ε, γίνεται λόγος ε, για το γεγονός ότι δεν εξαερώνεται το ποτόμα. Αυτό είναι εντελώς λανθασμένο και γελίο θα μπορούσα να πω τη στιγμή που ε, μπορούμε να μιλήσουμε και σε επίπεδο εκατοστολίτρων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί να μιλάμε για τη σύσταση του γάλατος των ε, μη αλκοολούχων ποτών και να μην μπορούμε να καλύψουμε τα αλκοολούχα. Την τελευταία φορά που το συζητήσαμε, πολλοί είπαν ότι η σύνθεση αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Ναι, αλλά τότε αλλάζει και, πολλές φορές αλλάζει και η σήμανση των υνοπνευματοδών. Ε, δεν χρειάζεται ε, απόλυτα, δεν χρειάζονται απόλυτα σωστά στοιχεία μέχρι το τελευταίο δηλαδή στοιχείο. Απλώς ε, χρειαζόμαστε στοιχεία σύνθεσης αυτών των αλκοολούχων. Θα υποβάλω τροπολογίες και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το απότερο μας μέλημα είναι να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Δεν ενοχλούμε κανέναν νομίζω. Τώρα η κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Γιούσο για τη δουλειά της, για αναθεώρηση του κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά δίδει στην Κομισιόν κάποια προνόμια, κάποιες εξουσίες που ξεπερνούν τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε κανονικά να έχει στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, η Κομισιόν έχει όλη την ευχέρεια να ρυθμίζει τις συνθήκες χορήγησης, τον έλεγχο, καθώς και την τροποποίηση της γεωγραφικής ζώνης ε, που αποδυναμώνει την αρχή αυτή των γραφικών ενδείξεων από την ουσία τους. Το παράδειγμα 3 του κανονισμού του 2008 που ε, αναφέρει όλους όλους τους γεωγραφικές ενδείξεις θα αντικατασταθεί από ένα ηλεκτρονικό μητρό και θα το ελέγχει μόνο η Κομισιόν χωρί κανένα δικαίωμα να ελέγξουν τα κράτη-μέλη αυτό το Μητρό. Επομένω, θα επαγρυπνούμε πάνω σε αυτό το θέμα που, κάτι άποψή μα, θα έπρεπε να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα καταθέσω, εννοείται, τροπολογίε για το θέμα αυτό. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε και άλλους βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν. Η κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Ιδίως γιατί εξέτασε και τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τι εξουσίες ε, μεταφέρουμε στην Επιτροπή. Στις πράξεις κατά εξουσιοδότηση έχει και δικαίωμα αρνηση στο Κοινοβούλιο. Πάντως, ε, πολύ σωστά το έλαβε υπόψη της η συγγήτρια. Επίσης, οι προτάσεις για αλλαγή του κανονισμού ε, βάση του κανονισμού για τα αλκοολούχα τα βάση του κανονισμού για τα ίδια τροφής ε, θεωρώ ότι είναι σωστό βήμα. Και θα ήθελα ε, να πω προς τους συναδέλφους ότι ήδη ο κανονισμός για τα τρόφιμα προβλέπει ότι πρέπει να αναγράφονται τα συστατικά. Και ο κλάδος τον οποίο τώρα η Επιτροπή ε, υποχρεώνει σε αυτορύθμιση, δεν αρκεί. Υπάρχει και ο κανονισμός ε, των ε, ειδών διατροφής Οπότε δεν χρειάζεται εμείς να προβλέψουμε εδώ κάτι καινούργιο. Ήδη προβλέπεται από τον κανονισμό για τα είδη διατροφής. Και για τα αλλεργιογόνα επίσης ο κανονισμός για τα είδη διατροφής περιλαμβάνει διατάξεις. σαν στο όνομα του προϊόντος ε, υπάρχει ο όρος ε, που είναι αντίστοιχο με το αλλεργιογόνο, δεν χρειάζεται να αναφερθεί επιπλέον. Αν είναι ε, κεράσι και κάποιος έχει αλλεργία στα κεράσια, είναι προφανής από τον τίτλο ή αν είναι λικέρ κεράσι αντιστοίχως. μου έκανε εντύπωση στην πρόταση της Επιτροπής ότι ορίζεται στο 37% ε, ο αλκοολομετρικός τίτλος ε, για τα προϊόντα που προέρχονται από Δημητριακά. Νομίζω ήταν 35% και θα πρέπει αυτό να παραμείνει. Ε, κάτι το οποίο λείπει είναι κάποιοι ορισμοί που θα είναι δεσμευτικοί, διότι τι θα πει ένωση, όταν μιλάμε για ένωση τι εννοούμε. Στο άρθρο 21 αναφέρεται αυτό και δεν είναι σαφές. Νομίζω ότι χρειάζεται ένας ξεκάθαρος ορισμός. Να μην μπορούμε να δώσουμε ό,τι ερμηνεία θέλουμε. Τι κριτήρια πρέπει να πληρούν αυτές οι ενώσεις. Επίσης, στο παράρτημα 1-2, ε, ο όρος απόσταξη, τι σημαίνει. Εννοούμε απλή απόσταξη και πολλαπλή απόσταξη. Θα πρέπει να είμαστε ακριβέστεροι λοιπόν για να υπάρχει και μεγαλύτερη ασφάλεια στον τομέα αυτό. Κάτι ακόμη που δεν καταλαβαίνω απολύτως αναφέρεται η εθιλική αλκοόλη από ίνο για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών. Η εθιλική αλκοόλη από μπύρα, παραδείγματος χάρη, τι διαφορά έχει γιατί και η μπύρα έχει συστατικά γεωργικής προέλευσης και θεωρώ σημαντικό και την θηλυκή αλκοόλη ε, για την πύρα να τη συμπεριλαμβάνουμε. γιατί να το επιτρέπουμε μόνο ε, στους ε, παραγωγούς είναι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συμπληρώσουμε. Για ορισμένα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει κάποιες ενδείξεις ε, να συμπληρωθούν. Αν γράφουμε την βότκα με V ή με W, πώς θα γράφουμε τη λέξη λικέρ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι γραφής των όρων αυτών, το είπε και η συγγήτρια και στην αγορά είναι γνωστά αυτά τα προϊόντα με συγκεκριμένες ε, με συγκεκριμένη ορθογραφική διατύπωση, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουν αυτά τα οποία είναι συνηθισμένα στην αγορά. Ένα άλλο ερώτημα είναι αν θα πρέπει να ε, συμπληρώνουμε και το άρωμα το οποίο έχει προσθεθεί σε ένα λικέρ. Λέμε πολλές φορές λικέρ καφέ ή λικέρ σοκολάτας ή το όνομα ενός φυτού το οποίο μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί γεντιανή παραδείγματο χάριν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους όρους που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν. Κάτι το οποίο ζητήθηκε και από άλλους συναδέλφους αφορά το σάκχαρο στα αποστάγματα ε, και εδώ θα πρέπει να έχουμε μια εναρμόνιση. Και όταν λέμε χωρίς προσθήκη σακχάρου, είναι κάτι το οποίο ε, εντάσσεται στις συζητήσεις και της Επιτροπής μας, ότι ε, η ζάχαρη παχαίνει. Ίσως θα μπορούσε λοιπόν ε, ένας τρόπος διαφήμισης να είναι ότι δεν, υπάρχει, δεν έχει προσταθεί καθόλου σάκχαρο σε ένα προϊόν. και εδώ υπάρχει ένα λικέρ με βάση το αυγό, χωρίς κρέμα. Στη δική μου περιφέρεια το φτιάχνουμε και με κρέμα και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε ε, να προσθέσουμε και την κρέμα στον ορισμό. Αλλά αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό για τον κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ντελάη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για αυτή την πρόταση. Τι λέει αυτή η πρόταση. Η πρόταση θέλει να εναρμονίσει τον τελευταίο γεωργικό κανονισμό τον 110 του 2008 και να τον ευθυγραμμίσει με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ας παραμείνουμε στα ουσιαστικά. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα με επενθυμίσω ότι πρόκειται για ένα τεχνικό κανονισμό και εμπορικό κανονισμό των αλκοολούχων ποτών και δεν μιλάμε για ένα κανονισμό που ασχολείται με την υγεία και προστασία των καταναλωτών απέναντι στο κίνδυνο που προέρχεται από την υπέρμετρη κατανάλωση υνοπνεύματος. Εάν συμφωνούμε επί του πλαισίου, επί του τι κάνουμε, του, του βασικού κανονισμού από το οποίο εγκύπτουμε, Πολλέ από τις συζητήσει και τα σχόλια τα οποία ακούσαμε σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα μας. Είναι εκτός θέματος. Να υπενθυμίσω ότι αυτός ο τομέας είναι ένα πολύ σημαντικό ε, οικονομικός πώ τομέας και εμπορικός πώ. Είναι ένας τομέας ο οποίος αντιπροσωπεύει, ίσως κάποιοι το βρουν αυτό περίεργο, αλλά είναι 10 δισεκατομμύρια εξαγωγών. 10 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγών. Και μιλάμε για χιλιάδε θέσει απασχόληση. Επομένω, προσοχή, προσοχή για το πώ προσεγγίζουμε αυτό το κείμενο, έτσι. Εγώ βλέπω διάφορα ερωτήματα προ την Κομισιόν κυρίω. Καταρχά, οι προτάσει που μα κάνει η Πιλάρ, η συγγήτρια, μου φαίνονται πολύ σωστέ. Η βασική μου Ερώτηση αφορά τη διαγραφή του παρατήματος 3 και την εφαρμογή αυτού του περίφημου ηλεκτρονικού μητρώου. Όχι ότι είναι αντίθετη με το μητρό αυτό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη γενικολογία γύρω από αυτό το μητρό και καλό θα ήταν η Κομισιόν να μας δώσει λίγα στοιχεία και διευκρινήσεις. Και τι δυνατότητες έχει να το τροποποιήσει μέσω εκτελεστικών πράξεων. Νομίζω ότι αυτές οι αρμοδιότητες δεν είναι και τόσο ευπρόσδεκτες. Έτσι. Δεύτερο ερωτηματικό που μου γεννάτε Μιλάμε για τη μετάφραση των ενδείξεων, των γεωγραφικών ενδείξεων, σε άλλα αλφάβητα, σε άλλες γλώσσες από αυτά που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. Μιλάμε κυρίως για το θέμα των εξαγωγών μας στις ε, χώρες της Ασίας. Η Κομισιόν στην πρότασή της δεν επιτρέπει τις μεταφράσεις. Τουλάχιστον ε, το επιτρέπει μόνο με μέσω ειδικών κατεξοδότηση πράξεων. Ε, πού είναι η απλούστευση εν αυτή περιπτώσει με την πρόταση αυτή τη Κομισιόν. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και συνεπείς ω προς το πώς θα συμπεριφερθούμε απέναντι στην πρόταση αυτή. Και εν πάση περιπτώσει, στην ε, Επιτροπή Γεωργίας, εγώ είμαι εισηγήτρια για αυτό το θέμα. Γι' αυτό θα προσέξω πάρα πολύ τις προτάσεις που θα κάνετε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ούτως ώστε να είμαστε συνεπείς πάνω σε αυτήν την πρόταση και να μην κάνουμε προτάσεις που κινούνται προς την μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, κατεύθυνση αποκλίνουσης μεταξύ τους δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Ντολάε. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν τον λόγο. Όχι, από ό,τι βλέπω. Άρα, από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, ο εκπρόσωπος Κομισιόν θα πάρει το λόγο. The Commission welcomes dialogue with Ευχαριστώ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της, του κανονισμού της Επιτροπής που έγινε το Δεκέμβριο του 2016. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κανονισμός 10-2008 για τα αλκοολούχα λειτουργήσε πολύ καλά στο παρελθόν και οδήγησε σε θέσεις εργασίας. Όμως εγκρίθηκε πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα αγροτικά με βάση τη συνθήκη. Άρα δεν θέλουμε να αλλάξουμε τους κανόνες, αλλά να ε, βελτιώσουμε το νομοθετικό κείμενο και να απλουστεύσουμε τις ε, επαχθές σε διαδικασίες των ε, γεωγραφικών ενδείξεων. Γι' αυτό λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις της κυρίας Αγιούζο που αποτελεί, κείμενο το οποίο αποτελεί μεγάλη βελτίωση του κειμένου σε σχέση με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Μιλάμε για έξι μήνες ελέγχου και αυτό το περιθώριο θα πρέπει να τύχει ε, περαιτέρω ανάλυσης και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα κράτη-μέλη ε, αποκλείουν τα πρόδειλα σφάλματα. Επίσης, θα πρέπει η Επιτροπή να κρίνει τη συμμόρφωση των ε, υπαρχουσών ε, γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται με βάση τον τρέχοντα κανονισμό και θα πρέπει να συνεχίσει. Βεβαίως, το νομικό μέσο ίσως να είναι διαφορετικό από, το, από του άρθρου 34. Η Επιτροπή θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, δεχόμαστε τις ε, τροπολογίες της ε, κυρίας ε, Ντελέη στην Άγκρη και Ντάντι στην Ίντα, που θα εξεταστούν περαιτέρω. Ε, όμως, έχουμε ορισμένες ανησυχίες σε σχέση με τα δεδομένα που προβάλλει η Επιτροπή Γεωργίας σε σχέση με τις προσμίξεις. Επίσης, η Επιτροπή Γεωργίας μίλησε για τις εθνικές διατάξεις που υπάρχουν για τις γεωγραφικές ενδείξεις και θα πρέπει να αλλάξουμε και τις αιτιολογικές σκέψεις για να μην υπάρχουν υπάρχουν ε, ε, λανθασμένες γεωγραφικές ενδείξεις, πλασματικές γεωγραφικές ενδείξεις στα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τα σύμβολα που ε, χρησιμοποιούνται θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο σε γεωγραφικές ενδείξεις, προστατευμένες γεωγραφικές ενδείξεις. Θα σας δώσουμε και περαιτέρω διασαφήσεις για αυτό το θέμα και θέλουμε να φτάσουμε σε ένα εξισορροπημένο πλαίσιο εξυγχρονισμού που να διέπει τα αλκοολούχα ποτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η κυρία Αγιούσο έχει το λόγο για, να, για σχόλια. Ευχαριστώ. Πριν κάνω τα σχόλιά μου, θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν, τη Γραμματεία, και την νομική υπηρεσία για τη βοήθεια που μου έδωσαν. Δεν το είπα πριν. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και πολύτιμη. Ευχαριστώ και τη, βοήθεια, τη βοηθό μου, τη Μάρτα, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ πάνω σε αυτήν την έκθεση. Σημείωσα όλα όσα είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Και αυτούς που συμφωνείτε και αυτούς που διαφωνείτε. Στην επόμενη συνεδρίαση θα συζητήσουμε και με τις τροπολογίες που είπατε, μπορούμε να βελτιώσουμε, ελπίζω, αυτή την έκθεση. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που υπόθηκαν, με αυτό που είπε η κυρία Σόμες για την μπύρα. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στο ενόπνευμα της μπύρας ή την μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και το σημαντικό είναι ότι όλα τα ενοπνεύματα που χρησιμοποιούνται στα αλκοολούχα ποτά να είναι Ινόπνευμα γεωργικής προέλευσης, αλκοόλ γεωργικής προέλευσης. Φυσικά μπορούμε να παρουσιάσουμε και τροπολογίες για το θέμα αυτό. Επίσης υπάρχουν θέματα, όπως ε, είπε και η κυρία Σόμες και άλλοι βουλευτές, δεν αφορούν αυτή την νομοθεσία, αυτό το νομοθέτημα, αφορούν την επισήμανση και άρα θα πρέπει να αριθμιστούν μέσα των άλλων νομοθετημάτων. Αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα, τεχνικός τεχνικό κείμενο και αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις των αρκολούχων ποτών. Αυτά σας ευχαριστώ όλους και είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά πάνω στο θέμα. Και εμείς ευχαριστούμε κυρία Γιούσο, σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τη συζήτηση. Για αυτό το θέμα έχουμε προθεσμία στις 7 Σεπτεμβρίου για τις τροπολογίες και ελπίζω να ψηφίσουμε στην ΕΜΒΗ στις 28 Νοεμβρίου. Κλείνουμε λοιπόν έτσι τη σημερινή μας συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει αύριο. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την ΤΕΒΕ και την ΕΚΟΝ, κοινή ανταλλαγή απόψεων. Σημαντικά θέματα. Θα σας δω αύριο το πρωί στις 9. Καλό σας βράδυ. Και μια και μιλούσαμε τόσο πολύ για ποτά, ε, να πιείτε και ένα ποτάκι. Σας ευχαριστώ.